Μα, εάν δεν έχετε αντίρρηση, εγκρίνεται η εντολή του. Επίση, οι γερμανικέ αρχέ μου είπαν ότι η διαδικασία άρση τη ασυλία του κυρίου Ούτο Βόικτ έχει ε, ανασταλεί από τον ε, εισαγγελέα του Σάρμπρουκ. Επομένω, η διαδικασία αυτή έχει έρθει στο πέρα τη. Από την ομάδα των Σοσιαλιστών και του ΕΛΚ έχω πάρει αιτήσει για διορισμού και αλλαγέ στη σύνθεση των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπιών. Θα προσαρτηθεί ο κατάλογο αυτό στα πρακτικά τη σημερινή ημέρα. Εάν δεν υπάρξει καμία αντίρρηση για την έκθεση των πρακτικών, θεωρούνται και αυτοί οι διορισμοί ότι έχουν εγκριθεί. Στην